Hello, everybody. Welcome to this press conference on the strengthening of the European border and coast guard. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου για την ενίσχυση της ε, υπηρεσίας για, τις, ε, για την προστασία των συνόρων και της εκτοφυλακής, την ε, γνωστή Frontex. Βγαίνουμε μόλις από την συζήτηση στην Ολομέλεια. Έχουμε την κυρία Μέτσολα, εισηγήτρια από το ΕΛΚ και τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο, υπεύθυνο για τη μετανάστευση και τα εσωτερικά. Η κυρία Μέτσουλα θα ξεκινήσει, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου για το Ευρωπαϊκό Σώμα Ακτοφυλακής, Φυλακής, Frontex και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ιδιαίτερος για την βοήθεια που μας προσφέρατε πριν να περάσω στην επισκόπηση των κύριων σημείων της πρότασης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αποτίσω φόρο τιμής στην μνήμη της Ντάφνε Καρουάνα Καλίτσια, της δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε ακριβώς πριν από 18 μήνες με τη χθεσινή ημερομηνία. Θα ήθελα λοιπόν να σου φορώ τιμή στη μνήμη της. Κανείς δεν φανταζόταν ίσως ότι θα μπορούσαμε όλη αυτή τη δουλειά να την ολοκληρώσουμε μέσα σε ένα εξάμεινο. Ε, πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο θα αλλάξει πολλά στη ζωή, την καθημερινή του κάθε Ευρωπαίου πολίτη και την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Χάρη στο νομοθέτημα αυτό λοιπόν μπορέσαμε ακριβώς να δώσουμε απαντήσεις στις ανησυχίες αυτές και να τις διασκεδάσουμε. Έχουμε υπόψη, λοιπόν, στις επιλογές μας τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαιοσύνης. Θέλουμε να είμαστε άτεγκτοι σε σχέση με αυτούς που προσπαθούν να παραβιάσουν τον νόμο, αλλά και να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τους πιο ευάλωτους Διατίθενται λοιπόν η απαραίτητη ανθρώπινη πόροι ώστε να επιτελεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό το έργο της η υπηρεσία με 10.000 νέους συνοριοφύλακες ή άλλο προσωπικό το οποίο στην επόμενη επταετία πρόκειται να προσληφθεί και αυτό πάντα μέσα σε μια ε, μέρη να παραμείνουμε ρεαλιστές και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μέχρι το τέλος του έτους και τα επόμενα έτη την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, ώστε η υπηρεσία να έχει την κατάλληλη επάνδρωση, αλλά και τα οικονομικά και τεχνικά μέσα που χρειάζεται, όχι μόνο τους ανθρώπινους πόρους. Θα πρέπει η υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της τα μέσα που χρειάζονται, ώστε να προσφέρει την αρρωγή της στα κράτη που την χρειάζονται και να καταπολεμήσει στα θέματα των επιστροφών βεβαίως να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, αλλά και να ε, υλοποιήσει ε, τα μέτρα που απαιτούνται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει η υπηρεσία να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε κάθε της δραστηριότητα και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να εγκαθιδρύσουμε ένα νέο φορέα, το παρατηρητήριο, με την υπηρεσία που θα μας επιτρέπει σε υψηλό επίπεδο να κάνουμε σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι δηλαδή πιο ρωμαλαία τώρα η διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχουμε εξασφαλίσει και ένα μηχανισμό υποβολής παραπώνων, όπως είχε προβληθεί πριν από τρία χρόνια, ένα στοιχείο θετικό. Έχουμε επίσης την ε, θέσπιση γραφείων ε, της υπηρεσίας σε τρίτα κράτη, ώστε να ενισχυθεί και η διάσταση της συνεργασίας με αυτά. Επίσης, στο κομμάτι που ενδεχομένως να μην είναι τόσο ελκυστική η υπηρεσία για τους υπαλλήλους, γιατί ο συντελεστής είναι σχετικά χαμηλός και έτσι δεν επιλέγεται ιδιαίτερα από υπαλλήλου που θα πηγαίνουν να δουλέψουν εκεί. Κάνουμε μία διόρθωση στο πλαίσιο του κανονισμού ε, δημοσίων υπαλλήλων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζει το θέμα αυτό. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί πολλούς έχει να κάνει με τις επιστροφές, με την υποχρέωση επιστροφών σε σχέση με τρίτα κράτη. Στη διακυβέρνηση πλειοψηφία σε κρατών μελών, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξασφαλίστηκε η πλειοψηφία. Και εδώ έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Στην πολιτική όμως των επιστροφών μπορέσαμε να ενισχύσουμε το σύστημα με ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό στην Ολομέλεια χάρη στην ε, συνεργασία μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε με τις λοιπές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μέτσολα. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότητες ευχαριστίες μου προς τη Ρομπέρτα Μέτσολα για την συνεχή άοκνη και ανεκτήμητη υποστήριξή της ε, στο θέμα αυτό. Ε, τα τελευταία χρόνια, μήνες, σε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκαν στενά και συντονισμένα για να καταλήξουν ε, σε ένα από τα πιο απτά και χρήσιμα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Εντολής. Μία πλήρως ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή. Αυτή είναι η σημερινή πρωτοβουλία και ελπίζω με την υπερψήφιση της σχετικής έκθεσης να αφήσουμε τη σχετική παρακαταθήκη σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από πέντε χρόνια διαχειριζόταν τα εξωτερικά τα σύνορα, δεν έχει καμία σχέση αυτός ο τρόπος με τη σημερινή κατάσταση διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Και με το πράσινο φως που θα δώσει σήμερα στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα από την τελική, οριστική έγκριση που θα γίνει από το Συμβούλιο της ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Και πολύ σύντομα αυτή, αυτό το ενισχυμένο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριακής και Ακτοφυλακής θα αρχίσει να αναπτύσσεται και πρόκειται ε, να φτάσει στο πλήρες δυναμικό των 10.000 ε, ατόμων μέχρι το 2027. Και θέλω να είμαι σαφής. Ε, δεν πρόκειται περί αναβολής. Δεν πρόκειται να περιμένουμε το 2027 για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Όχι, γιατί ήδη α, από τώρα, το 2021, το επιχειρησιακό προσωπικό θα αρχίσει να επεκτείνεται, να αυξάνεται. Γιατί πρόκειται μια σταθερή και σταδιακή διαδικασία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ήδη θα ενισχυθούν τα διάφορα γραφεία σύνδεσης ε, και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Και ε, το θέμα είναι ότι η επιχείρηση, εκτός από το μόνο προσωπικό, θα έχει και μέλη με εκτελεστικές εξουσίες για τη διεξαγωγή των, α, ε, της εξωτερικής διαχείρισης των συνόρων και της επιχείρησης επιστροφών. Και αυτό θα αρχίσει από την πρώτη μέρα εφαρμογής και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις επιστροφών, τα κράτη-μέλη χρήζουν περισσότερη υποστήριξη. Οπότε η ενισχυμένη ε, Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή θα μπορεί να τους επικουρήσει, να επικουρήσει τα κράτη-μέλη. Και μάλιστα τώρα οριστικοποιούμε τις συμφωνίες ε, για το καθεστώς με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και επίσης ε, προσβλέπω το συντομότερο δυνατό ο οργανισμός αυτός ε, να συνάψει σχετικές συμφωνίες και με χώρες πέραν της άμεσης γειτονίας μας. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να ε, αναχαιτήσουμε την παράτυπη μετανάστευση πριν φτάσει ήδη στα εξωτερικά μας σύνορα. Επίσης, θεωρώ ότι ε, θα μπορέσουμε να συστήσουμε και γραφεία επαφή στα κρατη και με τις εξωκοινωτικές χώρες ε, μετά την υιοθέτηση και του καθεστώτο, για να έχουμε και μια επιμελητιακή υποστήριξη των δραστηριοτήτων και να εξασφαλίσουμε μια εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του Οργανισμού Συνοριακή και Ακτοφυλακή. Και αν κάποιο αφισβητεί την προστιθέμενη αξία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση της μετανάστευσης και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, θα ήθελα να τον παραπέμψω, αν κάποιος έχει αφιβολή σε αυτή την ε, ε, συμφωνία και το επίτευγμα ορόσημο. Γιατί αν κάτι καταλάβαμε τελευταία πενταετία είναι ότι καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Και αυτός είναι, είναι και ο γενοσυργός λόγος ε, της σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριακής και Ακτοφυλακής. Όλοι συνειδητοποίησαν την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού σώματος και ενίσχυσης ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματο. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Εκτοφυλακή δεν μπορεί από μόνη τη να επιλύσει όλα τα ζητήματα. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε και το τελικό πράσινο φω, ώστε όλε ε, οι πληροφορίε ε, στο ενισχυμένο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών για αυτά τα θέματα να είναι διαλειτουργικέ. Και αν μια κόκκινη σημαία εμφανιστεί για κάποιον που φτάνει σε πέρασμα συνόρων, όχι μόνο θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό το άτομο από το να εισέλθει και να περάσει τα σύνορα, αλλά θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε αυτό το άτομο να εισχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Γιατί όλα τα, όλα τα συστήματα θα βλέπουν αυτή την κόκκινη σημαία λόγω της διαλειτουργικότητας της βάσης δεδομένων και οποιοδήποτε ε, θα περνάει τα εξωτερικά μας σύνορα θα ελέγχεται συστηματικά. Επίσης, να κοιτάξουμε λίγο τη γενικότερη εικόνα και την προέλευση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Και γι' αυτό από κοινού και συνολικά έχουμε αναβαθμίσει τη συνεργασία μας με πολλές ε, εξοκοινωτικές χώρες, μη ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα ήδη δρεύουμε τους καρπούς αυτής της συνεργασίας γιατί σταδιακά και κάθε χρόνο μειώνονται οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών. Και ενώπιση των ευρωεκλογών θα πρέπει να δείξουμε και στους Ευρωπαίους πολίτες ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τον προβληματισμό τους και ότι προσφέρουμε απτές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων λύσεων. Μια καλύτερη διαχείριση και καλύτερη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων είναι ο εξίσου σημαντικές για να προασπίσουμε και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χώρου Σέγγεν και των ελεύθερων μετακινήσεων. Ε, που είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες ε, που είναι ιδιαίτερα προσφυλής στους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι δείχνουμε σήμερα πόσο μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο έργο παράγει. Και θα ήθελα και πάλι να ξαναευχαριστήσω ε, την Ρομπέρτα Μέτσολα για τις εργόδεις προσπάθειές της, για την προσήλωση και τον ενθουσιασμό της ε, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά τα κατάφερε. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σαλβατορελούσο από την Άνσα και θα ήθελα να κάνω ερώτηση και προς, την, ε, προς τον Επίτροπο και προς την Συγκεκριά. Στην Ιταλία αυτή την ε, μεταρρύθμιση την έχουν επικρίνει οι δυνάμεις που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών. Τι θα απαντούσατε σε, αυτό τον, ε, σε αυτήν την επίκριση. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για να ακούσουμε και να απαντήσουμε ομού. Καλώ σας προχωρήσουμε με αυτήν. Κυρία Μέτσολα, ευχαριστώ πολύ. Όντως το ζήτημα αυτό το προέβαλαν αρκετοί οι περισσότεροι των εκπροσώπων των κρατών μελών εμείς καταστήσαμε σαφές ότι παραπέμπουμε στην αρχή της επικουρικότητας, ότι υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις εξουσίες και την αρμοδιότητα χρήσης όπλων από εκπροσώπους των δυνάμεων αυτών στο επίπεδο των κρατών μελών, στην επικράτεια των κρατών μελών και εν τέλει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις αλλά και οι ρόλοι αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη-μέλη αναλόγως δεν αλλάζουν. Παραμένουν όσοι έχουν. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος της δικής μας ε, στόχευσης με την αναθεώρηση. Θέλαμε να καταστήσουμε σαφές αυτό και βεβαίως θέλαμε να εξασφαλίσουμε για την υπηρεσία τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικών επιχειρήσεων και ανάπτυξης προσωπικού πιο αποτελεσματική στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό χρειάστηκε να το διευκρινίσουμε και το πράξαμε στο κείμενο. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι και το θυμό μας ότι ήταν εξ αρχής ένα από τα μελήματα των ε, κρατών μελών, των περισσότερων τουλάχιστον, ε, στο βαθ, σε ποιο βαθμό θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την εθνική κυριαρχία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εξασφαλίζεται απολύτω η εθνική κυριαρχία δεν χωρεί καμιά αμφιβολία. Δεν μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσει τη υπηρεσία χωρί συνένεση, θέλω να το καταστήσω το σαφέ. συνένεση των κρατών μελών ή και τη τρίτη χώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε όντως να καθοδηγήσει την υπηρεσία ως προς την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης επί τη βάση λειτουργικού σχεδίου που θα έχει συμφωνήσει η υπηρεσία με το εν λόγω κράτος μέλος. Επιπλέον και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπηρεσία μπορεί να παρεμβαίνει με εκτελεστικές εξουσίες σε τρίτες χώρες μόνο και επαναλαμβάνω μόνο επί τη βάση διεθνούς συμφωνίας που θα έχει το τρίτο κράτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λεγόμενες status agreements. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. Καλημέρα σας. Αμήνης Σέρα από τις Βρυξέλλες 2. Μία ερώτηση για την πραγματικότητα. Δηλαδή όλα αυτά εξαρτώνται από την υιοθέτηση ενός ε, ε, χρηματοδοτικού πλαισίου που θα εξασφαλίσει τους σπόρους για αυτές τις προσλήψεις, έτσι δεν είναι. Και μία άλλη ερώτηση θα ακούσουμε πριν απαντήσουν οι καλεσμένοι ή όχι. Την κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Η ε, κυρία Μετσόλα, αν κατάλαβα καλά, Ρωτήσατε για τα δημοσιονομικά μέτρα και πώς θα χρηματοδοτηθεί ο οργανισμός. Θα δούμε, γιατί η αρχική πρόταση προέβλεπε νωρίτερη προθεσμία. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούσε για την ανάπτυξη του προσωπικού μέχρι το 2021. Τώρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, υπάρχει μια παράταση μέχρι το 2027. Οπότε, η... τα χρηματοδοτικά μέσα θα εξαρτηθούν από τον αριθμό του προσωπικού και την κατανομή που θα γίνει σε αυτή την επταετία με τις διάφορες κατηγορίες που θα αναπτυχθούν. Αυτό που θα μπορούσα ίσως να προσθέσω είναι ότι μοιράσαμε τον αριθμό των 10.000 ατόμων τρόπο ώστε να μην έχουμε μια φέμαξη προσωπικού από τους εθνικούς φορείς, αλλά ταυτόχρονα ε, μεριμνήσαμε ότι σε περίπτωση κρίσης να έχουμε δυνατότητα ανάπτυξης και ταχείας αντίδρασης ε, στα εξωτερικά σύνορα, αν παραστεί ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στο δημοσιονομικό σκέλος. Και αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη από την αρχή να εξασφαλιστεί. Ε, φυσικά θα εξασφαλίσουμε τον απαραίτητο προϋπολογισμό για τον οργανισμό και ήδη προβλέπεται αύξηση τη συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Οργανισμό Συνοριακή και Εκτοφυλακή σε σχέση με την αρχική πρόταση που είχε προβλεφθεί στην πρόταση για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια σταδιακή μεν ομαλή δε ε, ανάπτυξη του μόνιμου σώματος συνοριακής και ακτοφυλακής από τις αρχές ήδη του 2027 και θέλουμε να λειτουργήσει εύρυθμα από την αρχή. Έχουμε 141 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2021 που συνιστά αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόταση. Τώρα εσείς εκεί στη μέση από την θα ήθελα να ρωτήσω ποιος αποφασίζει πού θα κατευθυνθούν οι μετανάστες. Δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Μπορεί να έχετε 10.000 άτομα προσωπικό, αλλά ποιος αποφασίζει η υπηρεσία στην πράξη. Πώς θα συμβεί αυτό. Κύριε Μετσόλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ήδη αυτό περιγράφεται στον τρόπο με τον οποίο ε, πραγματοποιούνται και οι τωρινές επιχειρήσεις είναι σαφές ε, και προσπαθούμε σε όλη την πορεία αυτή να εξασφαλίσουμε την ε, τήρηση του εθνικού δικαίου και η απόφαση σε σχέση με την... Ε, και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας και του κράτους μέλους θα συνεχίζεται. Σε σχέση με την αρχική πρόταση που είχαμε ε, την προσδοκία πως τα κράτη-μέλη θα προσέφεραν περισσότερο προσωπικό και δεν εξασφαλίστηκε αυτό, προσπαθώντας να περιορίσει τις ροές στα εξωτερικά σύνορα η υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Και ως εκπρόσωπος της ομάδας επαφής για το άσυλο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορώ να σας πω ότι θα θέλαμε να είχαμε στα προηγούμενα χρόνια πιο συγκεκριμένε αποφάσεις από το Συμβούλιο για την ε, υλοποίηση των λεγόμενων μηχανισμών αλληλεγγύης. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε εξασφαλίσει συμφωνία έτσι ώστε συγκεκριμένες αποφάσεις να λαμβάνονται άπαξ και κάποιος γίνει δεκτός στο επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι τύχη θα έχει η υποδοχή του, το αίτημα ασύλου, η περαιτέρω κατανομή. Όλα αυτά όμως έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο επίπεδο Συμβουλίου και δυστυχώς είμαστε εδώ στη τελευταία μας σύνοδο πριν από τις ευρωεκλογέ με εντολή και ήμουν εγώ συντάκτρια της αρχικής ολιστικής έκθεσης για την ε, ε, μετανάστευση στην οποία εντοπιζόταν η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών για τη μετανάστευση και εμείς εδώ έχουμε προχωρήσει αλλά έχουμε περιέλθει σε αδέξοδο σε επίπεδο συμβουλίου σε κάθε επίπεδο και έτσι σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα και έτσι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όχι μόνο σε μέτρα ε, ασφαλείας αλλά και σε μέτρα αλληλεγγύης να μπορέσει κάποια στιγμή η Ευρώπη να συμφωνήσει γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ερώτηση προς τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Πέρυσι το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα για τη χορήγηση ανθρωπιστικών θεωρήσεων και μέχρι τα τέλη Μαρτίου όφιλε να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αποδέχεται την πρόταση ε, και θα καταθέσει νομοθετική πρόταση ή όχι. Τελικά τι έγινε, ποια ήταν η αντίδραση, η επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις α, ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ο κύριος Αβραμόπουλος. We are seeing Το βλέπουμε αυτό στα πλαίσια της επανεγκατάστασης. Ε, λάβαμε την επιστολή με κάποιες ερωτήσεις και σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε. Since the votes are starting at 5 p.m. Ναι, θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ την συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε την κυρία Μέτσολα και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και σας ευχαριστώ όλους.